Opening our joint committee meeting. Και τώρα αγαπητοί συνάδελφοι κυρίσω την έναρξη της συνεδριάσεως μας της κοινή με την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών. Με χαρά λοιπόν καλωσορίζω τον συνάδελφο και συμπρόεδρο από την Επιτροπή των Πολιτικών Ελευθεριών. Πρώτο θέμα έγκριση της ημερής διάταξης. Έχετε παρατηρήσεις. Εγκρίνεται. Δύο ανακοινώσει Προέδρου, εγώ πάντως δεν έχω. Α, όχι, πρέπει να ανακοινώσω ότι θα έρθει στο Στρασβούργο η Επίτροπος Γιώουροβα, Δευτέρα, 15 Μαΐου, στη συνεδρίαση. Θα την υποδεχθούμε με μεγάλη χαρά. Περβάνς, θέλεις το λόγο. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ η δεύτερη ψηφοφορία απόρριψης που κατά πάσα πιθανότητα θα προκύψει από την ε, ε, μεικτή συνεδρίαση για τον κατάλογο αυτών. Είναι ένα σαφές μήνυμα πιστεύω προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πρέπει να εκφράσουμε και τη λύπη μας για το ότι δεν υπήρξε ποτέ ευκαιρία να συζητηθεί αυτή η πρόταση απόρριψης ε, στην εκδοχή Τη της κοινή συνεδριάσεω των δύο επιτροπών και με την ευκαιρία αυτής της ψηφοφορίας θέλω να επισημάνω με απόλυτη σαφήνεια τι είναι αυτό το οποίο απορρίπτουμε εκ μέρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής. Ένα κατάλογο χωρών κινδύνου Αφγανιστάν, Βοσνία, ε, Συρία, Ουγγάντα, Λάος, Παντμάτου, στη δεύτερη κατηγορία Ιράν, τρίτη κατηγορία Βόρεια Κορέα μετά την πρώτη μας απόρριψη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απλώς την Γουιάννα που την είχε στον αρχικό κατάλογο την αντικαθιστά με την Αιθιοπία στον ε, νεότερο. Ε, αυτό νομίζω πρέπει να το καταστήσουμε πολύ το σαφές ότι δεν είναι δυνατόν πλέον και εν τέλει χαίρομαι που η Επίτροπος δέχθηκε μια ανταλλαγή απόψεων με τους βουλευτές κατόπιν όλων όσων έχουν διαμειφθεί είναι πολύ σημαντικό και στην Ολομέλεια, στην ψηφοφορία μας αλλά και μετά την ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο οι δυο μας επιτροπές να διατηρήσουν την ε, πίεση που ασκείται απορρίπτοντας την πρόταση της Επιτροπής. Ο κύριος Φέρμπερ, με χαρά μπορώ να πω ότι συμφωνώ απολύτως με τα όσα είπες μεν, αφετέρου δε πρέπει και η Λίμπε να έχει, περιθώριο, να έχει στο περιθώριο των εργασιών της, στο πλαίσιο των εργασιών της και των χρονοδιαγραμμά τη αυτά τα θέματα, γιατί όπως έχουμε προβλέψει εμείς στη σχετική συνεδρία, πρέπει να έχει το χρόνο και η Λίμπε να το πράξει για να έχει και τη διερμηνία και όλα αυτά. Θα έρθει στο Στρασβούργο η κυρία Γιώροβα και φαντάζομαι ότι με την ίδια, τουλάχιστον με την ίδια χαρά, με αυτή που εκδηλώνουμε σήμερα, θα μπορέσουμε να δείξουμε απερίφραστα και ξεκάθαρα στην Επίτροπο Γιώροβα τι εννοούμε και τι θέλουμε. Θέλει κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Σημείο 3 ψηφοφορία και ευχαριστώ τη δεξιά πλευρά πτέρυγα για την υποστήριξη και ξεκινώ με μια επαλήθευση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Πρώτα με μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε αν δουλεύουν και αν υπάρχει κανένας περισεβούμενος. Ε, ε, μεταξύ των ψηφιζόντων. 15 μας λοιπόν. Για πατήστε οποιοδήποτε κουμπί. Προς το παρόν μόνο επαλήθευση κάνουμε του συστήματος. Ψηφίσαν όλοι. Έχουμε Ζατκόπ, Λάμπερτς, μην είναι και πολλοί οι σοσιαλιστές από πιο περισσότεροι ή οι πράσινοι αντίστοιχα. Περισσότεροι από ό,τι πρέπει άλλο θέμα αυτό. Εντάξει, δοκιμαστική ψηφοφορία ολοκληρώθηκε. Παράγραφος πρώτη υπέρ. Ηλεκτρονικά τα θέλετε όλα. Δεν ήθιστε στην ΕΚΟΝ, αλλά εάν θε το θέλει η ΛΥΜΠΕ. Ναι, μου λέει ο πρόεδρος της ΛΥΜΠΕ. Για να ικανοποιηθούν λοιπόν και οι συνάδελφοι της ΛΥΜΠΕ, Άρχεται η ψηφοφορία, παράγραφος πρώτη, ψηφίσατε όλοι, πέρας, εγκρίνεται. Δεύτερη παράγραφος, δεύτερη και μέχρι τέταρτη. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία πρώτη, τροπολογία δεύτερη, ταυτόσημες. Τις ψηφίζουμε. Α, όχι. Τεολογικό εδάφιο 6. Ψηφίσατε όλοι. 1 έως 6 ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 6 α. Τροπολογίες 1 και 2. Ταυτόσημες. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. και εγκρίνεται αιτιολογικό εδάφιο αρχικό κείμενο 7 και 8 ψηφίσατε όλοι πέρας εγκρίνεται A έως G, Z, Z, αιτιολογικές σκέψεις, αρχικό κείμενο, on block, ψηφίσατε όλοι, πέρας και εγκρίνεται. 8, αιτιολογική σκέψη, συγγνώμη, H, Ητά ε, ψηφίσατε όλοι πέρασε της ψηφοφορίας Φίλιπ μάλιστα δύο πρόσθετοι υπέρ επομένως 47 κατά 48 υπέρ άρα εγκρίνεται να ψηφίσουμε και το αρχικό κείμενο ένα λεπτό όμως αν, μπορούτε, αν μπορείτε να μου δώσετε μια εικόνα προς τους συναδέλφους, αγαπητοί φίλοι, γιατί με, σας κρύβανε, σας έκρυβε η κάμερα, δεν σας έδειχνε. Καταψηφίσατε. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό. Κατέλα, κατάλαβαν όλοι ότι αν ε, ο πρόεδρος δεν είναι ενήμερος ότι δεν έχετε την κάρτα μαζί σας, είναι δύσκολο να σας υπολογίσει στον, ε, στο αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Το έχετε αντιληφθεί. Λοιπόν, προτείνω το εξή. Θα κάνουμε για άλλη μια φορά τον, την καταμέτρηση. Τροπολογία 3. Καταρχάς ποιος δεν έχει κάρτα. Βάιτσέκερ Λάμπερτς. Εσείς έχετε κάρτα τώρα. Έχετε κάρτα. Καλά. Κα... Ξαναψηφίζουμε τροπολογία 3. Άρχεται. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απερίφθη. 49 κατά. 48 υπέρ. Αρχικό κείμενο. Αρχής ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και εγκρίνεται. Ψηφοφορία τροπολογία 4, αρχίζει ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας, Βάιστσέκερ κατά, Λάμπερτς κατά, απόρριπτα λοιπόν 45 κατά, 44 υπέρ. Γιώτα ή Άι, αρχικό κείμενο, αρχίζει ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται J, τροπολογία 5, αρχίζει η ψηφοφορία, ψήφισαν όλοι, πέρας. Εγκρίνεται, από ό,τι βλέπω, άρα δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε το αρχικό κείμενο. 6 σε τμήματα. Όπως έχει ζητήσει η ομάδα Σοσιαλιστών Δημοκρατών, ξεκινώ με το πρώτο τμήμα, αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. και έχει εγκριθεί. Στο επόμενο τμήμα, αρχής προφορία, ψήφισαν όλοι, πέρας. Και απορρίπτεται. Το κείμενο λοιπόν όπως ψηφίστηκε και τροποποιήθηκε ονομαστικά και αρχίζει η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι ο Φάουν Βάιτσέκερ υπέρ, ο Λάμπερτ υπέρ επίσης. Ναι, το χρειαζόμαστε μια κυριονομαστική ψηφοφορία, ε, πρέπει να το καταγράψουμε στα πρακτικά. Πέρ τη ψηφοφορίας και είναι σαφέ ότι εγκρίνεται η πρόταση. Σας ευχαριστώ θερμά. Κάτι άλλο έχετε, εγώ προσωπικός. Όχι, τα λέμε στο Στρασβούργο με την Επίτροπο Γιώργο. Καλό σα βράδυ.